μεταφερθούν όλε οι παρεμβάσει στον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτ και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα αυτό στην Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.